αντιμετωπίζουν. Η ε, είπατε εκπρόσωπο ε, βεβαίω συνεχίζει να, είναι, να έχει δεσμευτεί ότι θα συνεχίσει τι ε, προσπάθειε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ αγαπητή Επίτροπε. Λάβαμε μια πρόταση ψηφίσματο από την Επιτροπή Ανάπτυξη συγκεκριμένα και με αυτή την ανακοίνωση κλείνει η συζήτηση για το θέμα αυτό και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα σήμερα από τις 12 το μεσημέρι και μετά. Επόμενο σημείο, αγαπητοί συνάδελφοι, στην μερσιά Διάταξη αφορά εκ νέου προφορικέ ερωτήσει την Επιτροπή. Με θέμα αυτή τη φορά το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την ξενοφοβία και την ομοφοβία. η Πράσινη, η Ευρωπαϊκή Νοτική Αριστερά, η Φιλελεύθερη, η Προοδευτική Συμμαχία Σοσιαλιστών Δημοκρατών έχουν καταθέσει προφορικές ερωτήσεις για το θέμα αυτό. Για να δω τον κατάλογο των ομιλητών. Λοιπόν, μάλιστα. Πρώτη θα λάβει το λόγο η κυρία Ουλρίκη Λούνατσεκ ως συντάκτρια προφορικής ερώτησης. Δύο λεπτά έχει για την παρέμβασή τη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, η Ρωσία είναι πολύ σημαντική χώρα για τι εξωτερικέ σχέσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μέλο του Συμβουλίου τη Ευρώπη και έχει συνυπογράψει τι ευρωπαϊκέ δηλώσει για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, θεωρητικά λοιπόν έχουμε κοινέ ευθύνε για την προστασία των προτύπων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των σχετικών προδιαγραφών σε όλη την Ήπειρο. Αυτό που βλέπω όμω να συμβαίνει τώρα είναι ένα τρομακτικό φαινόμενο και μια κλιμάκωση τη βία κατά ορισμένων ομάδων του πληθυσμού μόλις ε, σήμερα το πρωί ε, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τους λεσβείς, τους ομοφιλόφιλους, τους αμφιφιλόφιλους, τους διαφιλικούς και τους φιλομεταβατικούς για ανθρώπους που θα μπορούσε να υποτεθεί ότι ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες. Πρόσφατα είχαμε δύο τουλάχιστον νόμους, έναν σε ομοσπονδιακό επίπεδο ε, του, της Αγίας Πετρούπολης ε, που απαγορεύει την διαφήμιση μη, παραδοσιακών σεξουαλικών πρακτικών προ ε, ανηλίκου. Αυτό σημαίνει ότι να μιλά κανεί για την ομοφιλοφιλία μπορεί να θεωρηθεί αδίκημα και μπορεί να φυλακιστεί ή μάλλον να πληρώσει πρόστιμο 22.000 ευρώ. Ε, για τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Ε, ένα κινηματογραφικό φεστιβάλ επίσης στην Αγία Πετρούπολη θεωρήθηκε ότι ήταν παράνομο. Δεν μπόρεσε να λάβει χώρα. Και κάτι ακόμη. Κάτι ακόμη που αποτελεί περίπτωση δικρατικής μεταχείρισης και κατά των σχετικών οργανώσεων. Υπάρχει ένας νόμος κατά τη χρηματοδότηση από το εξωτερικό. Δηλαδή, οποιοδήποτε ακτιβιστή μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το εξωτερικό θεωρείται κατάσκοπο ή ξένο πράκτορα. Αυτό που ουσιαστικά όμω παρακολουθούμε και κατασκοπεύουμε είναι πώ αντιμετωπίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα η Ρωσία. Μιλάμε για προπαγάνδα σε σχέση με την διάδοση μη παραδοσιακών σεξουαλικών πρακτικών προ ανηλίκου. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Πριν από εκατοντάδε χρόνια ε, πολύ γνωστοί Ρώσοι, όπως ο κύριος Τσαϊκόφσκι, ο μεγάλος, ε, ο Τσάρος Πέτρος. Ήταν γνωστό ότι είχαν ομοφιλοφιλικές σχέσεις και ότι ήταν ομοφιλόφιλοι. Τι θέλει ακριβώς λοιπόν η Δούμα με ένα τέτοιο νόμο, τι, η Δούμα, ε, τι επιδιώκει. Να αυξήσει την βία και να εντείνει την διακριτική μεταχείριση κατά των ομάδων αυτού του πληθυσμού. Κύριε Επίτροπε, λοιπόν, ε, το ερώτημα απευθύνεται προ εσά και προ το Συμβούλιο που δυστυχώ απουσιάζει. Τι κάνετε για να διασφαλίσετε ότι τα διαφελικά δικαιώματα προστατεύονται στη Ρωσία. Πρέπει να είμαστε πιο σαφείς και να δείξουμε πυγμή ε, στα θέματα αυτά. Τι κάνουμε με τους ανθρώπους αυτούς που είναι θύματα ταπείνωσης, που βιάζονται. Όταν οι άλλοι τους λένε δεν είστε άνθρωποι. Δεν είστε ανθρώπινα όντα. Ξέρουμε ότι έχουμε σοβαρά προβλήματα με αυτό του είδου τη βία κατά των ε, λεσβιών, των ομοφυλοφίλων, των αμφιλοφίλων, των διαφελικών και των φιλομεταβατικών. Τι θα κάνουμε λοιπόν ώστε στις ε, σχέσεις μας να ληφθεί υπόψη το θέμα αυτό και να κάνουμε κάτι. Σας ευχαριστώ Λορίκη Για δύο λεπτά ο συγητής ο Ντε Ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι προφανές ότι η θέση των ε, ε, ομοφιλοφίλων στην ε, Ρωσία είναι όλο και πιο δυσχερής. Βλέπουμε πάρα πολλά βίντεο στο YouTube με ανθρώπους που εξευτελίζονται λόγω της σεξουαλικής τους προτίμησης. Υπόκειται σε βία και όλα αυτά τα κρούσματα συμβαίνουν και σε άλλα κράτη και σε, άλλα κράτη, και σε κράτη-μέλη της Ένωσης. Οι περισσότερες για τι περισσότερες περιπτώσει, ε, τα κράτη-μέλη θα λάβουν κάποια μέτρα, είναι πιο εύκολο για τα θέματα να φτάσουν στο δικαστήριο, ε, δίνουν ε, εντολέ στι στις αστυνομικές αρχέ αρχές να αντιμετωπίσουν τέτοια κρούσματα, αλλά στη Ρωσία τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Οι αρχές κάνουν μάλλον το αντίθετο. Έχουν αυτό το, την νομοθεσία για την, για την προπαγάνδα και βλέπετε ανθρώπου στο YouTube ε, που ε, δείχνουν με χαρά τα, τα μαρτύρια που περνάνε. Ε, μας ζητούν λοιπόν να μην αντιδρούμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Εμείς θα πρέπει να ακούσουμε τους ανθρώπους στη Ρωσία όμως και ταυτόχρονα οι ίδιες οργανώσεις γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να βοηθηθούν από μόνες τους, χρειάζονται βοήθεια εξωτερική. Αυτό προφανώς δυσχεραίνει τα πράγματα. Γι' αυτό ένας αριθμός συναδέλφων, ε, μεταξύ των οποίων και ο υποφαινόμενος, έχουν λάβει πραγματικά απίστευτες απαντήσεις ε, σε ερωτήματα που έχουμε θέσει. Έχουμε στείλει επιστολές και στον ε, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχουν πολλά λόγια, αλλά δεν υπάρχουν πολλές πράξεις. Ακούμε ότι η ύπατη εκπρόσωπος λέει ότι πρέπει να δώσουμε υποστήριξη. Ε, ναι, αλλά αν απογορεύεται η υποστήριξη πώς θα τη δώσουμε. Πρέπει να προχωρήσουμε παρακάτω. Ας πούμε στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Θα πρέπει, λέμε, να πάρουμε μέτρα για να καταδείξουμε τα όσα γίνονται στη Ρωσία. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε, δεν μπορούμε να συνάψουμε μια συμφωνία. Και στρέφομαι σε εσά, κύριε Επίτροπε, έτσι ώστε να υπάρξει μια καλύτερη προσέγγιση για τα θύματα. Να παραδεχτούν ότι είναι θύματα τα οποία διώκονται στη Ρωσία λόγω των προτιμήσεών τους. Δεν μπορούμε λοιπόν να κάνουμε περισσότερα. Η Κομισιόν δεν μπορεί να μας εξηγήσει περισσότερο τι ακριβώς θα κάνει έτσι ώστε να γίνουν τα λόγια πράξη. Σας ευχαριστώ κύριε Ντεγιόγκ. Κανονικά τώρα ω συντάκτρια προφητική ερώτηση θα πρέπει να λάβει το λόγο η κυρία Κριστίνα Ογιουλάν, την οποία όμω δεν βλέπω ούτε στο δρανό τη ούτε γενικότερα στην αίθουσα. Γι' αυτό θα δώσω το λόγο στον κύριο Μάικλ Κάσμαν, που έχει δυόμιση λεπτά στη διάθεσή του. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, κυρία Επιτροπέ, είναι πολύ ενδιαφέρον που ο νόμος αυτός στη Ρωσία εφαρμόστηκε από το 2006, αλλά την ευθύνη την αναλαμβάνει ε, η κυβέρνηση, δεν την αναλαμβάνει η κυβέρνηση που ε, πρότεινε το νόμο αυτό το 1997 και ανέλαβε το 1998 Ο Σέξπιρ μας έχει δείξει με τα έργα του ότι πολλές φορές ε, το κακό ε, ξεπερνάει τη ζωή αυτών που το προκάλεσαν και φαίνεται και στα κόκαλα στους τάφους τους. Ο νόμος λοιπόν προτάθηκε το 97, να, ε, εγκρίθηκε το 98 και άρχισε να ισχύει από το 2006. Αλλά υπάρχει και ένας νόμος κατά της κατασκοπίας πλέον. Εδώ μιλάμε για καταπίεση όχι μόνο κατά των ΛΟΑΤ και των μη κυβερνητικών οργανώσεων που τους εκπροσωπούν, αλλά και για άλλους υπερασπιστές τέτοιων ομάδων μειονοτικών και υπόλοιπων ομάδων του πληθυσμού. Ε, εννέα οργανώσεις αυτή τη στιγμή ε, διώκονται. 18 έχουν λάβει επίσημη εντολή έχουν κατηγορηθεί μάλλον για κατασκοπία και περισσότερες από 30 έχουν λάβει προειδοποίησεις να μην παραβιάζουν τον νόμο. Αυτοί οι νομικοί περιορισμοί συνοδεύονται από εκφοβισμό, από παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών των ανθρώπων και από δίωξη των ε, ανθρώπων που συμμετέχουν σε αυτές τις ονέσεις. Ποιέ είναι αυτές οι παραδοσιακές της Ρωσίας. Ε, πώς επερασπίζεται τις εθνοτικές ε, μειονότητες, ε, τους μετανάστες και τους ΛΟΑΔ. Οι νόμοι αυτοί δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές ρωσικές αξίες. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα ατσάλινο χέρι το οποίο με δικτατορικό τρόπο ε, χρεώνει στη σιωπή ε, και την ε, απομόνωση αυτές τις ομάδες του πληθυσμού. Η Ρωσία πρέπει να σεβαστεί τι υποχρεώσει τη για τα ανθρώπινα δικαιώματα συμπεριλαμβανόμενε τη Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το θέμα αυτό. Αλλά κυρία Επίτροπε, πρέπει και εσεί και το Σώμα των Επιτρόπων και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση να κάνετε δύο πράγματα τουλάχιστον. Πρώτα απ' όλα να παρακολουθείτε τι εξελίξει στη Ρωσία, όχι μόνο με τι κατευθυντήρε γραμμέ για του ΛΟΑΔ, αλλά με συνεχή διοργάνωση ε, διαλόγου σε διμερέ επίπεδο και σε συνόδου κορυφή και με συνεχεί συνομιλίε, αλλά ίσω και με του χειμερινού Ολυμπιακού Αγώνε, με τέτοιε αφορμέ. Θα πρέπει να συζητήσει βελτιώσετε επίσης το καθεστώς θεωρήσεων, ε, κυρία Επίτροπε, ε, με την ε, Ρωσική Ομοσπονδία. Δεν πρέπει να τους κάνουμε δώρα στην καμπούρα αυτών που έχουν πέσει θύματα εκμετάλλευσης και βίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Μάκη, Κυρία Επίτροπε, η σειρά σας τώρα για να απαντήσετε στο συντάξει των προφορικών ερωτήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Γνωρίζω ότι πολλές φορές τον τελευταίο μήνα έχει εκφράσει το σώμα την ανησυχία του για το θέμα αυτό. Και εμείς συμμεριζόμαστε την ανησυχία των Ευρωβουλευτών για την κατάσταση των ανθρωπινών δικαιωμάτων στην Ρωσία. Καταρχάς να σας διαβεβαιώσω ότι οι ανησυχία που εκφράσατε ε, έχουν ληφθεί υπόψη με αποφασιστικότητα, γιατί από την αρχή η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέστησε σαφέ ότι η Ρωσία θα πρέπει να σέβεται τι διεθνεί τη δεσμεύσει και να αγωνιστεί για ένα σύστημα που θα βασίζεται πλήρω στο κράτο δικαίου, το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε μια όλο και πιο δημοκρατική κοινωνία. Και πολλέ φορέ επισημαίνουμε την ε, ασυμβατότητα μεταξύ κάποιων νομοθετημάτων ε, για τι διαδηλώσει, για τη λασφημία, για την ελθοτυπία, για την ε, φιλοφιλική προπαγάνδα, πώς τη λένε, τον έλεγχο του διαδικτύου κτλ. κτλ. Όλα αυτά τα θέματα που αναφέρατε ε, μας να αναφέρουμε δύο ε, νομοθετήματα. Το ένα αφορά τη, τους ξένους ε, πράκτορες και έναν άλλο νόμο που αφορά τα παιδιά και τους ε, ανηλίκους. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακούσαμε αυτά που λέτε και την Πρώτα απ' όλα, Συνεχίζουμε έντονε διπλωματικέ προσπάθειε να εκφράσουμε τι ανησυχίε μα ό,τι αφορά την εφαρμογή των νομοθετημάτων αυτών. Η ΕΠΑΤΗ εκπρόσωπο δημοσία αντιδρά όποτε, κάθε φορά που εγκρίνονται ή ε, δημοσιοποιούνται τέτοιοι νόμοι. Επίση, συστηματικά θέτουμε τα ζητήματα αυτά σε όλε τι συνομιλίε που έχουμε με του Ρώσου ομολόγου μα σε ό,τι αφορά το, λόγο που, το νόμο που απαγορεύει την ομοφιλοφιλική προπαγάνδα, όπως λέμε. Λέμε ότι στιγματίζει κάποιες ομάδες πληθυσμού και παροτρύνει, οθεί σε βία. Επίσης, διαβουλεύσεις και για ανθρώπινα δικαιώματα και σε άλλους πολιτικούς διάλογους. Τα θέτουμε αυτά τα ζητήματα. Εγώ στις τακτικές επαφές που έχω με τις ρωσικές αρχές, ιδίως με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Εσωτερικών, επανειλημμένως θέτω και στη Μόσχα το θέμα αυτό, αλλά και εδώ στις Βρυξέλλες και αλλού. Επίσης, στη Μόσχα Είχαμε ειδικέ ε, ανταλλαγέ ε, και για το Προεργικό Συμβούλιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, που είναι και στην πρώτη γραμμή ε, για τι προτάσει τροποποίηση αυτών των νομοθετημάτων. Και στο Κατερίνα στη Σύνοδο Κορυφή τον Ιούνιο. Η εκπρόσωπο, αντιπρόεδρο Άστον, έχει τονίσει συγκεκριμένε ανησυχίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί συρρυκνούται ο χώρο τη κοινωνία των πολιτών, οδηγώντα τη Ρωσία σε λάθο κατεύθυνση. Πρέπει λοιπόν να είναι καλύτερε οι διαβλέψει για τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα πρέπει οι σχετικέ διαβλέψει να γίνονται στην Μόσχα με συμμετοχή των Ρώσων Υπουργών. Ο επόμενο γύρο συνομιλών προβλέπεται για το επόμενο έτο. Επίση, δραστηριοποιούμεθα και στο πολυμερέ επίπεδο. Πρόσφατα καλέσαμε το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στι 17 ε, Σεπτεμβρίου συγκεκριμένα ε, στην ε, διάσκεψη του ΟΗΕ να θέσει ε, υπόψη της Ρωσίας τις ανησυχίες μας για αυτά τα δύο νομοθετήματα και να ζητήσει από τη Ρωσική Ομοσπονδία να κάνει ό,τι μπορεί ώστε να είναι σεβαστά τα βασικά δικαιώματα, η ελευθερία έκφρασης, να είναι πιο αποφασιστική στη δράση της, να υπάρχει ανοχή απέναντι σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας. Τα ίδια λέμε και στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον ε, ασε και ελπίζουμε ότι τελικά θα υλοποιηθεί ε, η νομοθεσία αυτή και αυτά τα οποία περιμένουμε και για το επόμενο έτος με την Επιτροπή της Βενετίας. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν πολλέ μη κυβερνητικέ οργανώσει και Ρωσική Ομοσπονδία με τα ανθρώπινα δικαιώματα και κινδυνεύουν, όπω η ε, Γκόλο, που είναι μια ε, οργάνωση παρατήρηση εκλογών που τη επιβλήθη πρόστιμο και έκλεισε. Άλλε οργανώσει δεν έχουν πάρει ε, χρηματοδότηση, ε, θεωρούνται ξένοι πράκτορε. Όλα αυτά ε, στόχο έχουν είτε να φημώσουν είτε να λογοκρίνουν μέσω εκφοβισμού, μέσω περικοπής της χρηματοδότησης όλες αυτές τις οργανώσεις. Παρ' όλα αυτά, εμεί πρέπει να βοηθήσουμε, να στηρίξουμε ε, τις οργανώσεις αυτές να συνεχίσουν το θεμητό τους έργο προστασία δημοσιογράφων, δικαιώματα μειονοτήτων, όλα αυτά συνιστούν ε, την ε, καθεδρής κράτου δικαίου στη Ρωσία. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις οργανώσεις κοινωνία των πολιτών και μέσω της πατσαρμοστία στη Ρωσία. Και στην περιοχή και στις Βρυξέλλες θα συνεχίσουμε να ε, έχουμε επαφέ και συνεργασία με τη ΜΚΟ. Ο ειδικό εκπρόσωπο για τα δικαιώματα, πολύ γνωστό σε εσά, ο Σταύρο Λαμπρινίδη, ε, με την κοινότητα των πολιτών, με του διάφορου αξιωματούχου, έχει στενή επαφή. Θα ταξιδέψει ε, τον ε, μήνα αυτό στη Ρωσία. Και βέβαια, πάντοτε θα τονίζουμε ότι είμαστε ανεξάρτητοι, δεν είμαστε ποτέ πράκτορες και στα τέλη Σεπτεμβρίου στην επισκέψη μας το είπαμε ε, και στην τελευταία Γενική Συνέλευση του Φόρουμ Κοινωνίας των Πολιτών Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας το είπαμε τη Δευτέρα και επίσης από τα κράτη-μέλη ε, παρακολουθούμε και το κατά πόσο είναι δίκαιο το δικαστικό σύστημα, αν απονέμεται σωστά η δικαιοσύνη, η διακριτική μεταχείριση των μειονοτήτων, ε, οι παραβιάσεις του κράτους δικαίου, δεν θα επηρεάσουν θετικά τις σχέσεις μας με τη Ρωσία. Δεν θα ενισχύσουν ε, ε, τις σχέσεις συνεργασίας μας. Πρέπει να το γνωρίζει αυτό η Ρωσία. Θα πρέπει λοιπόν να σεβαστεί τις δεσμεύσεις της και να σεβαστεί και τις αρχές του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εμείς βέβαια θα στηρίξουμε τη Ρωσία. Είναι γείτονα, είναι στρατηγικός εταίρος, αλλά με ειλικρινή και επικοδομητικό τρόπο στο πλαίσιο του διαλόγου μας. Ευχαριστώ. ευχαριστώ πολύ. Κυρία Επίτροπε, Περνάμε στους ε, εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Εκ μέρου του ΕΛΚΑ έχει το λόγο ο κύριος Κρίστοφ Λίσεκ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, πριν μιλήσω για τη Ρωσία θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ένα πολύ θλιβερό ε, νέο που μόλις έλαβα τώρα το πρωί ο κύριος Μάρτενς πέθανε. Πέθανε ε, πριν λίγα λεπτά και θα ήθελα να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στην ε, οικογένειά του. Ε, πριν ψηφίσουμε θα ήθελα να τιμήσουμε, Πρόεδρε, αυτόν τον πολύ καλό συνάδελφο και ένα εξαιρετικό Ευρωπαίο. Τώρα, για τη Ρωσία. Χάρηκα πολύ που άκουσα τα όσα είπε η Επίτροπος μόνο να τα υποστηρίξω μπορώ, να τα συνυπογράψω. Ε, συμφωνώ απολύτως με κάθε σας λέξη. Θα μπορούσα να κλείσω εδώ, μάλιστα. Χαίρομαι και που η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σύνολό τη είναι τόσο δραστήρη στην ε, όλη διαδικασία έτσι ώστε να αλλάξει αυτό το πολύ περίεργο νομοθετικό κείμενο. Είναι είναι πολύ περίεργο, είναι απαράδεκτο τον 21ο αιώνα να υπάρχουν τέτοιε νομοθεσίε. Και θα πρέπει βεβαίω και εμεί να έρθουμε σε επαφή με τι δικέ μα κυβερνήσει, τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και εκεί να πιέσουμε για την Ρωσία. Αυτός ο νόμος είναι σκανδαλώδης και δεν θα πρέπει να έχει το βάρος μόνο η Επίτροπος ή η Υπατή Εκπρόσωπος για να δράσουν. Ε, οποιοςδήποτε, όλοι οι Πρωθυπουργοί, οι Υπουργοί Εξωτερικών, όταν έρχονται σε επαφή με τη Ρωσία θα πρέπει να λένε ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε μια κατάσταση όπου υπάρχουν τέτοιες νομοθεσίες. Ενισχύει όπου τα βασικά δικαιώματα καταπατώνται. Ευχαριστούμε, συνάδελφε. Να ζητήσω από τους σοσιαλιστές να πάρουν τώρα το λόγο. Ο κύριος Ενρίκε Γκερέρο θα μιλήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Επίτροπο. Θα ήθελα και εγώ να δείξω την αλληλεγγύη μου στην οικογένεια του Βίλφρεντ Μάρτεν που μόλις μάθαμε ότι απεβίωσε. Βεβαίως δεν ανήκε στην ίδια πολιτική ομάδα με εμένα αλλά η πολιτική μου ομάδα και η δική του ε, μοιράζονται κοινέ αρχές και αυτό ε, έχει σχέση και με το θέμα που, ζητούμε, που συζητούμε σήμερα. Σεβασμό στις ε, ανθρώπινες, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην ανθρώπινη υπόσταση. Ε, όταν ε, παραβιάζουμε την ε, ανθρώπινη υπόσταση το κάνουμε με πολλούς τρόπους και για πολλούς λόγους γιατί δεν δείχνουμε σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών. Ένα από αυτά τα δικαιώματα είναι η ελεύθερη επιλογή του καθενός για την σεξουαλική του, το σεξουαλικό του προσανατολισμό. Ζητούμε λοιπόν από τη Ρωσία να σεβαστεί το κράτος δικαίου και κάνοντα αυτό δεν μιλούμε μόνο για την υπεράσπιση των, ανθρωπι... ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, μια μειονότητα ή μια πλειοψηφία. μιλούμε για την προστασία των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των ε, ανθρώπων. Είναι μια ανθρω... Η ανθρώπινη υπόσταση διακυβεύεται όταν άνθρωποι καταπατούν τα δικαιώματα των συμπολιτών του. Οπότε υποστηρίζω απολύτω τα όσα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον... και ο κύριο Λαμπριανίδη. Ε, η Ρωσία όντω είναι μια μεγάλη ε, χώρα εταίρος και έχουμε ε, διαφόρων ειδών σχέσεις με τη Ρωσία το θέμα δεν είναι μόνο οικονομικό ούτε θέμα ενέργειας είναι οι αξίες που ε, υπερασπιζόμαστε στην Ευρώπη και που διακυβεύονται τώρα εκ μέρους των πρασίνων η κυρία Ινφελτ ευχαριστώ πρόεδρε κυρία Επίτροπε Βλέπουμε ότι το Συμβούλιο αποσιάζει, όπως συνήθως, πολύ ωραία. Τέλο πάντων, πολλά υπόθηκαν για όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη Ρωσία. Όλοι ανησυχούν ιδιαίτερω για τι πρόσφατε εξελίξει. Νομίζω ότι ο συνδυασμός αυτών των συγκυριών είναι πιο ενισχυτικός. Υπάρχει ο νόμος κατά της ομάδας των ΛΟΑΔ. Υπάρχει ένας ακόμη νόμος ο οποίος θέλει να εκφοβήσει και να περιορίσει τις με κυβερνητικές οργανώσεις. Αλλά πάνω απ' όλα έχει ο πρώην πράκτορας της ΚΑΚΕΜΠΕ, ο κύριος Πούτιν, αναγγείλει την ε, υλοποίηση ενός προγράμματος για μαζική παρακολούθηση των πολιτών για σκοπούς εθνικής ασφάλειας. Νομίζω ότι αυτό το πρόγραμμα θα το επιτρέψει να παρακολουθεί τους ανθρώπους, να τους εκφοβήσει και στην ουσία να τους κάνει να σιωπήσουν και να τους φημώσει. Μιλάμε για ένα νέο είδος λογοκρισίας. Θα πρέπει να είμαστε λοιπόν πολύ πιο επίμονοι εδώ. Να μην συζητάμε μόνο για διάλογο με τον κύριο Πούτιν. Νομίζω ότι δεν έχει καμία απολύτω σημασία για τον κύριο Πούτιν ο διάλογος. Άλλα πρέπει να κάνουμε και θέλω να κάνω εδώ κάποια σχόλια. Πρώτα απ' όλα τη στάση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Δεν είναι δική μας δουλειά, αλλά πραγματικά ε, σοκάρομαι και πραγματικά τρομάζω από την απαράδεκτη στάση τους. Ε, πώς δείχνουν την υποστήριξή τους τις... Ε, ε, ομάδες των ΛΟΑΔ και των ε, μη κυβερνητικών οργανώσεων λένε ότι θα ήταν ανάμειξη στα πολιτικά της Ρωσίας. Μα πώς γίνεται αυτό, ο κύριος Πούτιν και η χώρα του είναι μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Πώς είναι πολιτική παρέμβαση το να ζητά κανείς να γίνει σεβαστός ο νόμος για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό δεν είναι πολιτική στάση στα πράγματα. Επίσης, θα έπρεπε να πω στην, Ευρωπαϊκή, στην Ολυμπιακή Επιτροπή και στα μέλη της ότι η σιωπή είναι και αυτό ένα μήνυμα εύγλωτο. Είναι ένα μήνυμα μήνυμα υποστήριξη προ τον κύριο Πούτιν. Ήθελα λοιπόν να καλέσω την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή να αναθεωρήσει και να μεταβάλει τη στάση τη. Εδώ, ω Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόκειται να προσχωρήσουμε στην ECHR. Ε, Δεν μπορούμε λοιπόν εδώ στην ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ να αποδυναμώνουμε τους κανόνες και τα πρότυπά της. Θα πρέπει να σκεφτούμε την αναστολή της ε, συμμετοχής της Ρωσίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Αυτό πρέπει να αρχίσει να συζητάτε ως προοπτική. Και να ρωτήσω και την Επίτροπο, τι θα γίνει με την απελευθερώση του καθεστώτος θεωρήσεων ε, ε, για τη Ρωσία. Πολλά ακούγονται, αλλά τίποτα δεν βλέπουμε να γίνεται στην πράξη. Συνάδελφοι, νομίζω ότι Ολοκληρώνοντα, μια τελική πρόταση αρκεί. Να δείξουμε τη στήριξή μα προ τι ομάδε του πληθυσμού, των ΛΟΑΔ και των μη κυβερνητικών οργανώσεων και με την ε, χρηματοδότηση, την ε, χρηματοδοτική μα υποστήριξη προ του ανθρώπου αυτού. Να αγνοήσουμε την απαγόρευση για τη χρηματοδότηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Μιλάμε εδώ για τι βασικότερε αρχέ και αξίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Εκ των Πρασίνων για 1,5 λεπτό έχει το λόγο Μαρία Κορνέλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ρωσία είναι ένας μεγάλος γείτονας, ο μεγάλος μας γείτονας και θα ήθελα να προσεγγίσει περισσότερο την Ένωση, παίρνει τα κινήσεις, ε, ε, εμπορικές σχέσεις σε όλες τις πτυχές όμως το καθεστώς την απομακρύνει τη Ρωσία αντίθετα αντί να την προσεγγίζει αυτή η προπαγάνδα κατά των ομοφιλοφίλων είναι ένα φρικτό ε, σημάδι που δείχνει καταστολή για όλα όσους δεν συμφωνούν με του κυρίου Πούτιν Επίσης, ό,τι αφορά ε, τις ε, μη κυβερνικές οργανώσεις που λαμβάνουν χρηματοδότηση από το εξωτερικό και θεωρούνται πλέον ξένοι πράκτορες με βάση τον νέο νόμο, αυτό και έχει επίσης φρικτές συνέπειες. Επίσης οι νεαροί ομοφιλόφιλοι απειλούνται, έχουν διωχθεί, έχουμε συνεχώς κρούσματα βίας κατά ατόμων ΛΟΑΔΑ. Ακτιβιστές ε, ε, φυλακίζονται, διώκονται. Πολλοί όμως θεωρούν ε, την κυβέρνηση Πούτιν φιλική, την κανονική κυβέρνηση. Στη χώρα μου, την Ολλανδία, φέτος Νοτάζουμε τα 400 χρόνια των δεσμών μας με τη Ρωσία και θα γίνουν του κόσμου εορταστικές εκδηλώσεις από εδώ και από εκεί. Αν και δεν βλέπω τόσο πολύ ένθερμη τη φιλία τον τελευταίο καιρό, πιστεύω ότι θα πρέπει ε, τις ρωσικές αρχές ε, να μην τις αντιμετωπίζουμε ως φίλους. Δεν είναι φίλοι μας, δεν είναι φίλοι των ανθρωπίνων, ε, μάλλον των αστικών δικαιωμάτων, ούτε και του ρωσικού λαού φίλοι δεν είναι. Είναι φίλοι μόνο του καθεστώτος και της δυναμής τους. Δεν μπορεί να υπάρξει περαιτέρω απελευθέρωση του εμπορίου του καθεστώτος θεωρήσεων χωρίς να υπάρχει μεγαλύτερο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των ατόμων λάθη δηλαδή, στη Ρωσία. Δεν μπορούμε να συναντώμεθα με ομολόγους μας από τη Ρωσία και να γιορτάζουμε εδώ τις σχέσεις μας και την ιστορία τη Ρωσία, εάν δεν ε, μένουμε και δεν τονίζουμε το ζήτημα των δικαιωμάτων όπω τη ελευθερία έκφραση. Και στο Συμβούλιο τη Ευρώπη θα πρέπει ε, να τεθεί αυτό το ζήτημα. Επίση θα πρέπει να αποφύγουμε να επιδεινωθεί η κατάσταση αυτή γιατί καθημερινά αυτό βλέπουμε. Πρέπει να στηρίξουμε το ρωσικό λαό αφού του εγκαταλείπει η κυβέρνησή του. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ κυρία Κορνέλσεν. Έχει τώρα το λόγο για ένα λεπτό ο Δόκτωρ Τάνοκ. Κύριε Πρόεδρε, από όλο το πολιτικό φάσμα πολύ ε, βλέπουμε, μάλλον παρατηρήσαμε με πολύ μεγάλη χαρά την κατάρρευση του σιδηρού παραπετάσματο στην ελευθερία του πρώην ε, Σοβιτικού Μπλοκ. Όμω ο κύριο Καρκόσκι 10 ε, χρόνια φυλακίστηκε, θύμα τη Εμπληκτική δικαιοσύνη και παραμένει στη φυλακή. Και λέω για αυτόν τον άνθρωπο γιατί δείχνει ότι έχουμε συνεχή παρακμή στην κατάσταση ανθρωπινών δικαιωμάτων και κράτο δικαίου στη Ρωσία που ουσιαστικά κηρύσσει ως εχθρού αυτούς οι οποίοι θέλουν να ζήσουν σε ειρήνη χωρίς να βλάπτουν κανένα. Οι μειονότητες, τα άτομα ΛΟΑΔ, εφίστανται ε, διαχείριση. Αυτό δεν περιορίζεται βέβαια μόνο στη Ρωσία, αλλά αν δει κανεί τη γλώσσα, τη ρητορική που ακούγεται στη Ρωσία αυτή τη στιγμή, δείχνουν να ξανανομιμοποιούν αυτή τη βία. Ε, και πρόσφατα πέρασε και από τη Δούμα αυτό το νομοθέτημα για την ομοφιλοφιλική ε, προπαγάνδα. Και προωθούν προωθούνται παραδοσιακέ οικογενειακέ αξίε, όπω λέμε. Αυτοί οι άνθρωποι για του οποίου μιλώ όμω δεν έχουν ίδια σε μια ελεύθερη δημοκρατική κοινωνία. Και υπάρχουν πολλοί οι οποίοι κάνουν ε, ζωντανή κόλαση τη ζωή αυτών των ανθρώπων. Ε, φημώνουν, κόβουν ε, τη δυνατότητα έκφραση τη ταυτότητα ορισμένων ομάδων. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πώ θέτει αυτά τα θεμελιώδη θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κράτου δικαίου στη Ρωσία. Άκουσα τι είπε η Επιτροπό Μάλστρομ και κανένα δεν αμφιβάλλει πόσο σημαντική είναι η πολιτική, οικονομική, στρατηγική σχέση, η σχέση ασφαλής με την Ρωσία. Πρέπει όμως να μιλήσουμε ε, ανοιχτά για αυτές τις διακρίσεις και για, αυτή, για αυτές τις ε, ταπεινώσεις που υφίστανται αυτές οι ομάδες. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Η ε, κυρία Κορνίλια Έρνστ τώρα έχει το λόγο εκ μέρου ε, τη Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά. Ευχαριστώ. Θυμάμαι κάποια είδηση που άκουσα στην ε, τηλεόραση για μια Ρωσίδα η οποία ήταν ε, στο ε, στάδιο και κρατούσε ένα πλακάτ για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης. Την έβρισαν, την χτύπησαν, ε, την έδιωξαν οι αστυνόμοι. Ε, Ήταν πραγματικά ε, πέσια κατάσταση. Η ομοφοβία είναι μια κατάσταση που δημιουργεί πάρα πολύ αρνητικέ συνέπειε στην Ρωσία. Θεωρούνται αυτοί οι άνθρωποι ανώμαλοι, άρρωστοι. Πρέπει λοιπόν επιγόντω αυτό το θέμα να το αντιμετωπίσουμε. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι παγκόσμια. Πρέπει να ισχύουν για όλου και πάντα και βεβαίω και πρέπει να ισχύουν στη Ρωσία. Χρειάζεται διάλογο λοιπόν γι' αυτό με τη Ρωσία, με κυρώσει. Δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Πρέπει να μιλήσουμε, να μιλήσουμε σοβαρά. Γι' αυτό υποστηρίζω την προσέγγιση της Επιτρόπου που πραγματικά πιστεύω ότι δουλεύει σκληρά, προσπαθεί να ανοίξει αυτή τη συζήτηση, ίσως να είναι και η μόνη που το κάνει και πραγματικά θυμώνω που το Συμβούλιο πάντα πάντα σε τέτοια θέματα και δεν παρεμβαίνει σε, σε τέτοια θέματα. Παρόλο που υπάρχουν ε, ε, χώρες που ε, έχουν περιπτώσεις ομοφοβίας. Κυρία Επίτροπε, συνεχίστε. Είναι πραγματικά εξαιρετική σημασία στο θέμα αυτό. Εγώ θέλω να ξαναπάω στην Ρωσία με ήσυχη τη συνείδησή μου, να πάω να κάνω διακοπές και πραγματικά θέλω να συνεχίσετε την προσπάθειά σας. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Έρνστα. Τελευταία παρέμβαση σε αυτό το γύρο. Είναι η παρέμβαση του κυρίου Στάτερ, του μη εγγεγραμμένου. Πρόεδρε, αυτό το κοινοβούλιο πριν από λίγες εβδομάδες έβλαβε ε, μία απόφαση για την ε, ε, μη παρέμβαση στα εσωτερικά θέματα των εταιρικών χωρών. Όλη η συζήτηση όμως δεν θεωρείται παρέμβαση στην, στα εσωτερικά της Ρωσίας. Το ίδιο αυτό κοινοβούλιο δεν κάνει τίποτα για χώρες όμως όπως η ε, Σαουδική Αραβία όπου κάθε, χώρα, ε, κάθε χρόνο κρεμνιούνται άνθρωποι λόγω της σεξουαλικής τους ε, προτίμησης. Στη Ρωσία δεν ε, υπάρχουν συγκρίσιμες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως υπάρχουν στην Τουρκία για παράδειγμα. Ε, νομίζω ότι θα χάσουμε την αξιοπιστία μας απέναντι στην ε, Ρωσία αν κάνουμε μια αντιρωσική συζήτηση. Και τα δύο νομοθετικά κείμενα που υποβρίσκονται εδώ υπό συζήτηση έχουν τύχει τη μεγαλύτερη υποστήριξη από του Ρώσου πολίτε. Και πρέπει να έχουμε την συμφωνία των ε, των Ρώσων πολιτών. Είναι θέμα εσωτερικό της Ρωσίας αυτό που μπορούν οι Ρώσοι να το ρυθμίσουν μόνοι τους. Πρέπει να δούμε λοιπόν ε, να, να μην θεωρηθεί η δική μας παρέμβαση ως παρέμβαση στα εσωτερικά της. Η Ρωσία μπορεί να κανονίσει μόνη της ε, τα θέματα αυτά. Οι Ρώσοι πολίτες όμως δεν είναι σαν, ε, σαν εμάς. Οι Ρώσοι πολίτες αυτή την συζήτηση την κάνουν πάρα πολύ χαλαρά κανένας δεν τους ε, τρομοκρατεί και πραγματικά ας αφήσουμε την ε, συζήτηση αυτή στους Ρώσους να την κάνουν. Μάλιστα. Να περάσουμε τώρα στους λοιπούς ομιλητές. Πρώτα απ' όλα για δύο λεπτά θα δώσω το λόγο στην κυρία Στριφλέρ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπο, αγαπητοί συνάδελφοι, από την έγκριση πολλών νόμων περιορίζουν τα ελευθερία έκφραση, ε, του συνέρχεστε, του συνεταιρίζεστε και ιδίω ε, αυτό ο νόμο για του ε, ξένου πράκτορε ή κατά τη προπαγάνδα, οι επιθέσει, η βία, τα φαινόμενα ξενοφοβία, ομοφοβία πολλαπλασιάζονται. Αγνοούνται, παραγνωρίζονται όλο και περισσότερο και κατάφορα τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία. Αυτός ο νόμος για την προπαγάνδα, την ομοφιλοφιλική, ε, αυξάνει τις διακρίσεις ε, που ήδη είναι πολύ έντονες στη Ρωσία κατά των ατόμων ΛΟΑΔ. Ε, Κρίνεται μέσα σε ένα πλαίσιο Τρομερή ε, απομόνωση ομοφιλοφοβία στη Ρωσία. Πρέπει να το καταδικάσουμε. Καθήκον μα είναι να συνεχίσουμε να ευαισθητοποιούμε τι ρωσικέ αρχέ για τι δραματικέ επιπτώσει των νόμων αυτών. Να του υπενθυμίσουμε ότι πρέπει να συνεχίσουν να σέβονται τι διεθνεί του δεσμεύσει. Είναι επιτακτική ανάγκη η Κάθριν Άστον, η Εκπρόσωπο και η ΕΕΔ να ε, έχουν έναν διάλογο ε, έντονο και συνεχή για αυτά τα θέματα και αυτές τις παρεμβάσεις. Ευχαριστώ Μισελ. Λέω πρόεδρος, για 1,5 λεπτό έχει το λόγο τώρα η κυρία Τζοάννα Σενίτσι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να ενδυναμώσει τις σχέσεις της με την ε, Ρωσία. Όμως θα πρέπει ταυτόχρονα να σεβόμαστε τι δημοκρατικέ αξίε και τα ανθρωπίνα δικαιώματα και έτσι ισχυριζόμαστε ότι κάνουμε. Ε, δεν μπορούμε λοιπόν να παραβλέπουμε το γεγονό ότι δεν σέβεται τι υποχρεώσει τη αυτέ η Ρωσία, έτσι όπω προκύπτουν από το εθνικό δίκαιο. Η σύμβαση Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα αλλά και Διεθνεί Συμβάσει για τα Δικαιώματα των Πολιτών ε, είναι κείμενα τα οποία η Ρωσία έχει δεσμευτεί να σέβεται. Εδώ μιλάμε για βίαιε επιθέσει κατά των πολιτών τη Ρωσία με το πρόσχημα της ε, των σεξουαλικών του προτιμήσεων. Η μεταχείριση των μη κυβερνητικών οργανώσεων, ο σχετικός νόμος που απαγορεύει την ε, δυνατότητα του συγκεντρώνεστε και του διαδηλώνει είναι ανησυχητική και Υπάρχουν ανησυχητικέ διώξει ε, κατά των δημοσιογράφων, των ακτιβιστών από ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ούτω καθεξής. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ούτω ή άλλω, υπήρξε μια έκθεση για, για το κράτο δικαίου και την προστασία του δικαίου στη Ρωσία. Οι δράσεις μας ως τώρα δεν έχουν φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Σε τελευταία λοιπόν, ε, ως τελευταία λύση θα πρέπει να προσπαθήσουμε να πείσουμε τις αρχές της Ρωσίας ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βελτιώνει και την εικόνα της Ρωσίας στο διεθνές προσκήνιο και κυρίως τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ συνάδελφε. Για ένα λεπτό τώρα έχει το λόγο ο κύριο Μπένιον. Δεν τον βλέπω στην αίθουσα. Ίσως να βγει και για λίγο. Να δώσω τώρα το λόγο λοιπόν για ένα λεπτό στον Άνταν Μπίλαν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, εδώ ο νόμος ε, της Ρωσίας για την ε, ξένη κατασκοπία ουσιαστικά καθιστά υποκείμενες ε, αδικήματα τουλάχιστον 300 ε, με κυβερνητικές οργανώσεις ε, με κυβερνητικέ οργανώσει που παρακολουθούν την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την προστασία του και το πώ εξελίσσεται το κάτω δικαίου στη Ρωσία. Η Γκόλου είναι μια ανθρωπιστική οργάνωση που παρακολουθεί εκλογέ και έχει υποστεί τι σοβαρότερε κυρώσει. Καταλαβαίνουμε τι επιπτώσει έχουν τέτοια φαινόμενα στο δημοκρατικό καθεστώ τη Ρωσία. Και καταλαβαίνουμε βεβαίως τι ενέργειες μπορεί να προβεί ο ρωσικός στρατός. Ήδη έχουν οργανωθεί στη Μόσχα ασκήσεις και επιδείξεις που θυμίζουν το σοβιετικό καθεστώς. Δεν μπορούμε να παραμένουμε αδρανείς μπροστά σε τέτοια φαινόμενα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Κούκαν τώρα έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ρωσία για πολλούς και διαφορετικούς λόγους βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής μας. Είναι πολύ πιθανό ούτε η χάρτα των Ολυμπιακών Αγώνων να μην γίνει σεβαστή και αυτό δείχνει μια κατάσταση, καταδεικνύει μια κατάσταση πολύ ανησυχητική. Η Ρωσία ασκεί καταστολή ε, στο εσωτερικό της ίδιας της χώρας και στις γειτονικές χώρες. Είναι πολύ ενισχυτικό το γεγονός ότι η πίεση ασκείται και ε, προς τα έξω αλλά και στο εσωτερικό. Ε, οι ρωσικές αρχές βάζουν στο στόχαστρο το, την κοινωνία των πολιτών και εκφοβίζουν τον πληθυσμό της χώρας και τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις αλλά και ξένους ε, πολίτες. Ο λεγόμενος νόμος κατά της προπαγάνδας εκφράζει ακριβώς την υποβάθμιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία τους τελευταίους μήνες. Αυτά δεν επιτρέπουν μόνο την άσκηση πίεσης, αλλά δίνουν και λαβές σε πολύ νοσηρέ ερμηνείε. Υπάρχουν ε, ομάδε του πληθυσμού που είναι πραγματικά ευάλωτε, αλλά αντιμετωπίζονται ω πολίτε δεύτερη κατηγορία. Επιπλέον, όταν η Ρωσία ε, ασκεί πίεση σε γειτονικέ χώρε όπω η Αρμενία, η Ουκρανία. ή τις χώρες της Βαλτικής. Ε, ασκείται πίεση και προς Ανατολάς και προς Δυσμάς. Ε, είδαμε προσφάτα εμπορικέ κυρώσεις κατά της Λιθουανίας. Δεν μπορούμε εδώ να παραμένουμε αδρανείς. Ε, πρέπει να εκφράσουμε τις αντιρρήσεις μας με τρόπο κατηγορηματικό και σαφή. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό το λόγο έχει ο συνάδελφος Ρέπου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι συνεπής στις σχέσεις που έχει με τη Ρωσία. Πρέπει να μιλούμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για την ε, εξέλιξη της δημοκρατίας. Είναι σημαντική η συνεργασία μας με τη Ρωσία, ωστόσο πρέπει να μας ενδιαφέρει και να μας ανησυχεί η κατάσταση του κράτους δικαίου και των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Δεν θα πρέπει να δεχόμαστε κατάφορες ε, παραβιάσεις της δημοκρατίας ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Αυτά τα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο είναι σοκαριστικά. Βλέπουμε επιθέσεις ε, βιαιότατες κατά των ε, ο ατόμων ε, ΛΟΑΔΕ και δεν είναι δυνατόν ε, να απειλούνται οργανώσεις οι οποίες καταγγέλουν τέτοια περιστατικά να απειλούνται λοιπόν ε, με διακοπή της χρηματοδότησής τους με αποκλεισμό. Όλα αυτά είναι σε αντίθεση με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει διεθνώς η Ρωσία. Η Ρωσία είναι ο μόνος υπεύθυνος που θα πρέπει να διορθώσει την κατάσταση. Μια ανοιχτή, ε, πολύμορφη κοινωνία είναι πλούτος για τη Ρωσία και γενικότερα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό έχει το λόγο ο κύριος Στρέιτσεκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα σας, κυρίε και κύριοι. Καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης ακούω πολύ προσεκτικά και όντως συμμερίζομαι αρκετά από τα επιχειρήματα και τα σχόλια των συναδέλφων. Αλλά θέλω να πω ότι κάτι που θα μπορούσε να έχει υποθεί, αλλά δεν το άκουσα. Ε, εγώ ε, ζούσα στην ε, κομμουνιστική Τσεχοσλοβακία και βεβαίως δεν έχω κανένα λόγο να υπερασπιστώ οτιδήποτε έχει να κάνει με την, Ευρωπαϊκή, με την Ρωσία. Συγγνώμη. Αλλά ε, η Ρωσία δεν είναι η Σοβιετική Ένωση, ε, δεν υπάρχει κομμουνισμός στη Ρωσία. Η Ρωσία δεν ε, εξασκεί τα, όσα, τα ίδια με τις ίδιες πρακτικές με αυτές που υπήρχαν πριν από 30-35 χρόνια. Ναι, είναι αλήθεια ότι η Ρωσία μπορεί να μην κινείται με το σωστό τρόπο προς την δημοκρατία. Μπορεί να είναι δύσκολος αυτός ο δρόμος, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει ε, πρόοδος σε σχέση με πριν από τόσα χρόνια. Πολλοί Ρώσοι είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι και ε, πιστεύουν σε συγκεκριμένες αξίες μπορεί να, ε, θεωρήσουν ότι είναι εξευτελιστικά τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούμε εμείς σήμερα εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Βάιντεν Χόλτσερ για 1,5 λεπτό. Δεν τον βλέπω στην αίθουσα. Παίρναμε λοιπόν στον τελευταίο για αυτό το γύρο παρεμβάσεων ομιλητή, τον αντιπρόεδρό μας Βλάσακ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, η αρνητική προσέγγιση από τι ε, ρωσικέ αρχέ προ τι μειονότητε και τι μη κυβερνητικέ οργανώσει αλλά και του ανεξάρτητου ε, δημοσιογράφου με τι πολιτικέ δολοφονίε και τη βία αποτελούν παραδείγματα που δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι δημοκρατικέ αρχέ στη Ρωσία δεν ε, γίνονται σεβαστέ. Αυτοί που θέλουν να τι υπερασπιστούν αντιμετωπίζουν βία και ψευδείς κατηγορίες και η ζωή τους πολλές φορές απειλείται. Γι' αυτό πρέπει να πούμε πολύ δυνατά ότι παρά τις προσπάθειες δεν έχουμε καταφέρει να αλλάξουμε την ρωσική στάση απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν έχουμε καταφέρει να βελτιώσουμε την άσχημη κατάσταση που επικρατεί. Τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά ε, μόνο στη θεωρία θεωρούνται πολύ σημαντικά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την ε, Ρωσία. Δεν θα επηρεάζουν δηλαδή τις ε, σχέσεις μας, ε, ας πούμε, τις εμπορικές. Επίσης, κάποια κράτη έχουν αλλάξει την εξωτερική τους πολιτική μετά από την πίεση της οικονομικής κρίσης και αρχίζουν να προτιμούν τις ε, εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία. Γι' αυτό πρέπει να επαναλάβουμε τα όσα λέμε και να συνεχίζουμε να επιτονίζουμε τη σημασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σας ευχαριστούμε κυρία Βλάσακ. Ε, περνάμε στους ε, ομιλητές που προσέλκυσαν την προσοχή του Πρόεδρου μέσω της διαδικασίας Catch the Τέσσερις στον αριθμό συγκεκριμένα. Ο πρώτος που θα λάβει το λόγο είναι μία συνάδελφος συγκεκριμένα, η κυρία Πέτροβιτς. Και Παρότι ζήτησε το λόγο όμως δεν τη βλέπω στην αίθουσα. Προσέλξε την προσοχή μας αλλά της... ήταν αρκετό αυτό μάλλον διότι αποχώρησε. Ο κύριος Ντόνσκης τώρα που είναι μέσα στην αίθουσα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, το παράδοξο της υπόθεσης είναι ότι αντί να εορτάζουμε την, αντί να εορτάζει η Ρωσία την, τη μεγάλη της ιστορία στην στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους μεγάλους εκπροσώπους της υπεράσπισης αυτών όπως ο Ζαχάροφ, ο Μπουκόφσκι και άλλοι ουσιαστικά μιλάμε για τα θηριωδίες που έκαναν άνθρωποι όπως ο Στάλιν και άλλοι ε, προσπαθούν δηλαδή να στιγματίσουν κρατήσουν σήμερα ανθρώπους της κοινότητας των ΛΟΑΔΑ, δημοσιογράφου κτλ. Η χώρα που έχει κάθε δικαίωμα να ε, εορτάζει την ε, μεγάλη της κληρονομιά στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ουσιαστικά ε, κατηγορείται από το, από το δικαστήριο για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παρόλο που υπάρχει το βραφείο Ζαχάροφ, το μεγαλύτερο βραβείο του 20ου αιώνα προσπαθούν να στιγματίσουν τους καλύτερους ε, της Ρωσίας και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να το δεχτούμε αυτό. Σας ευχαριστώ Λεωνίδας. Ο κύριος Πολ Μέρφιτ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η νέα νομοθεσία τη Ρωσία που απαγορεύει την προώθηση των μη παραδοσιακών σεξουαλικών σχέσεων έχει ε, δημιουργήσει ένα κύμα αντιδράσεων ε, και βία κατά τον, ε, τον ΛΟΑΔ. Βεβαίω, αυτό ήταν και ο σκοπό τη νομοθεσία, να στείλει ένα σαφέ μήνυμα ότι η ε, το κράτος ε, ε, δικαιολογεί τη βία κατά των ομοφιλοφίλων. Κατηγορούνται, τους μιλούν με απέσια στους επιθετικούς προσδιορισμούς, τους βασανίζουν, δέρνονται. Δική μου φίλη στην Ρωσία, ας πούμε, ο Ιγκορ Γιάσεν από την, από την σοσιαλιστική αντίσταση, το σχετικό, τη σχετική ένωση, έχουν πάρει μέρος σε διαδηλώσεις, έχουν, τους έχουν για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτή η νέα νομοθεσία λοιπόν ε, μειώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και μάλιστα θα γίνει ε, η απαγόρευση του Gay Pride στην, ε, στη Μόσχα. Άνθρωποι έχουν φτάσει να κάνουν ε, απεργία πείνας ε, και τα μέλη της ε, ΛΟΑΔ είναι αυτά που τελικά πλήττονται. Όλοι όσοι θέλουν να υπερασπιστούν τα δικαιώματα των εργαζομένων, τα δικαιώματα των ομοφιλοφίλων, τα δικαιώματα των ανθρώπων πρέπει να λάβουν τη σωστή θέση. Ευχαριστώ πολύ. τελευταίο ομιλητή, ο κύριο Μπρόν, για αυτό το γύρο. Επίτροπε, είπατε ότι θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός για το δίκαιο και τους νόμους στη Ρωσία. Όμως, εδώ δεν αντιμετωπίζουμε τις παραβιάσεις του, πραγματικού δικαίου, του κανονικού δικαίου. Ε, ακούσαμε στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών την ενδεχόμενη καταδίκη ανθρώπων που κατηγορούνται στην Ελλάδα για φρικτές δολοφονίες ε, και οι οποίοι μπορεί να έχουν καταδικαστεί προτού εκδικαστεί η υπόθεσή τους. Πώς μιλάμε λοιπόν για, την, ε, για το σεβασμό του κράτους δικαίου στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Ας το δουν αυτό πρώτα τα ίδια τα κράτη-μέλη για τους εαυτούς τους. Η Ρωσία είναι ένα κυρίαρχο κράτος που μπορεί να κάνει ό,τι νομίζει. Εάν όντως παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, αυτό θα ήταν κάτι το... Ε, ποινικά κολλά, θα ήταν κάτι το που θα μπορούσε να επισύρει κατηγορίες. Αλλά Είμαι βέβαιος ότι πολλοί βουλευτές εδώ μιλούν ειλικρινά και από καρδιάς. Όμω η συζήτηση αυτή υποκρύπτει προτεραιότητες που δεν έχει καμία σχέση με τι σεξουαλικέ ελευθερίε, την ελευθερία της έκφραση, αλλά με την εξωτερική πολιτική τη Ρωσίας κατά βάθο. Ευχαριστώ. Ε, Μάλιστα. Ολοκληρώσαμε με το γύρο αυτό, και θα δώσω το λόγο στην ε, Επίτροπο, η οποία με την δευτερολογία της θα κλείσει τη συζήτηση για το θέμα αυτό. Σεσίλια, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αποτίσω φόρο τιμής στον κύριο σε έναν μεγάλο Ευρωπαίο, φυσικά τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του, στους φίλους του. Ήταν λίγο ζωφερή συζήτηση, αλλά θα σα δώσω μια καλή είδηση. Υπήρχαν έλεγχοι 100% σε φορτηγά από τη Λιθουανία που είχαν επιβληθεί από τη Ρωσία. Αυτοί οι έλεγχοι ανεστάλησαν. Αυτό είναι μια καλή είδηση. Βέβαια, διατηρεί το αποκλεισμό των γαλακτοκομικών προϊόντων. Αυτή ήταν η καλή είδηση. Τώρα έχουμε στι κακέ ειδήσει. Ε, όλο και περισσότερε ε, έχουμε ανησυχίε. Ε, Κουζέγκο, τη Μηγορία την Τρίτη. Ε, ψυχιατρικός εγκλισμός. Αυτό μας θυμίζει κακές ε, αναμνήσεις από το παρελθόν. Επίσης, η επιστολή της κυρίας ε, Κουνικών από το συγκρότημα Pussy Riot, που, Pussy Riot η οποία είναι και σε απεργία πείνας που κυκλοφόρησε. Ζητούμε λοιπόν να μπορεί να τη δει η οικογένειά της, η δικηγόρη τη και να ε, βελτιωθούν οι συνθήκε κρατησή τη. Τα τελευταία είναι για την Greenpeace επίσης μας έχουν ανησυχήσει και στις Βρυξέλλες και στη Μόσχα και με την Greenpeace και με τα κράτη-μέλη και τα πρεσβεία και τα Είμαστε σε συνεχείς επαφές Προ το παρόν. Ε, ακολουθούμε προξενική προσέγγιση. Θέλουμε τα 30 άτομα που συνελήφθησαν να αφαιθούν ελεύθεροι. Το ίδιο και το, το σκάφος. Δεν θέλουμε να γίνεται λόγο σε καμία περίπτωση για ε, πειρατεία. Σε ό,τι αφορά την απελευθέρωση των θεωρήσεων, θέλω να σας πω ότι έχουμε τέσσερα ε, πεδία διαπραγμάτευση. Ένα από αυτά είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτό είναι και το πεδίο στο οποίο έχουμε σημειώσει τη λιγότερη πρόοδο. Και συνεχίζουμε να θέτουμε το θέμα σε όλου του διαλόγου, σε όλα τα επίπεδα, υπουργικό και άλλα επίπεδα με τι ρωσικέ αρχέ. Λυπούμε που δεν ε, είχα απαντήσει στο ερώτημά σα τώρα. Ε, να πω ότι με εξέπληξε η συνένεση εδώ στο Κοινοβούλιο Όλους μας ανησυχεί άκρος η κατάσταση, ιδίως με αυτά τα δύο νομοθετήματα, αλλά και για άλλα θέματα. Στην εισαγωγική μου ομιλία σας έκανα μια μακροσκελή αναφορά ε, στις δράσεις ε, της ΕΕ εκπροσώπου και της Επιτροπής εν γέννη. Συνεχίζουμε να αξιοποιούμε όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για να καταδικάζουμε τα κακό και να ζητούμε αλλαγέ. Βλέπω και ακούω την πλήρη σας υποστήριξη και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είμαι σίγουρη ότι θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό γιατί δεν φαίνεται ότι σύντομα θα έχουμε κάποιες ριζικές αλλαγές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για τη σημαντικότητα αυτή συζήτηση. Πρόεδρος, με την παρέμβαση της κυρίας Μάλστρομ ολοκληρώθηκε η συζήτηση για το θέμα αυτό. Ψήφισμα δεν υπάρχει, επομένως δεν θα υπάρξει ψηφοφορία. Επί του θέματος ολοκληρώνεται λοιπόν η συζήτηση και περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Jó reggelt kívánok! A következő napirendi pontunk a Macmillan Scott jelentés. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η αιτήσια έκθεση του Edward Macmillan Scott για τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2012. Ο κύριος Macmillan Scott δυστυχώς δεν είναι εδώ σήμερα μαζί μας. Οπότε η κυρία Ματσόνη.